Members, if we could restart, that would be... Να αρχίσουμε, συνάδελφοι. Αν καθίστε αυτό θα βοηθήσει και έτσι να υπάρχει το χρονικό περιθώριο. I'm sure we had more people than this just now. Okay, thank you. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης αφορά την επιλογή των ε, προεδρευόντων στο δευτεροβάθμιο όργανο του Ευρωπαϊκού ε, Οργανισμού για την Πνευματική Ιδιοκτησία. Και πρόκειται να βρεθεί κάποιος από το Συμβούλιο, από κάποιον κατάλογο υποψηφίων. Στις 22 Δεκάτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έστειλε το κατάλογο των υποψηφίων. Δύο από αυτοί, οι φιναλίστ Αντρε Πόλμαν και Αλεχάνδρα Κονσάλε Φερνάντεθ και είπαμε ότι πριν αποφασίσει το Συμβούλιο πρόκειται να ε, προβεί ο υποψήφιος, ο κάθε υποψήφιος σε κάποια δήλωση και γι' αυτό τους έχουμε εδώ ε, και καλέσαμε τέλος πάντων ε, αυτόν που επελέγει από το Συμβούλιο, δηλαδή την κυρία Βιρτζίνια Μέλγκαρ, η γραμματεία μας έχει οργανώσει μια διανομή του βιογραφικού των υποψηφίων και θα έχετε χρόνο 10 λεπτών για να προβείτε στη ε, δήλωσή σας και να απαντήσετε τις τυχόν ερωτήσεις στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να αρχίσω για αυτή την σύντομη δήλωση. Πρώτα πρώτα να αυτοσυστηθώ πέραν του βιογραφικού που σας έχει διανεμηθεί. Είμαι Γαλλίδα αλλά γεννήθηκα στη Νότια Αμερική σε μια μικρή χώρα την Ουρουγουάη. Όμως, στα 17 ήρθα στην Ευρώπη και σπούδασα νομικά και εγκληματολογία στο Παρίσι. Έγινα το 82 δικαστής στη Γαλλία. Μετά από δύο χρόνια εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Κατόπιν διορίστηκα στις Βερσαλίες εισαγγελέα και μετακινήθηκα σε ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου υπηρέτησα πέντε χρόνια και το 1991 προσλήφθηκα στην νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ε, εθνικός εμπειρογνώμων ε, όπου με έστειλε η γαλλική κυβέρνηση. Επομένως ε, είχα το προνόμιο και την τύχη να βρεθώ εκεί τρία χρόνια σε αυτή την σαρπαστική περίοδο πριν ε, ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Δούλεψα για εναρμόνιση εσωτερική αγορά το 1994. Ήμουν ο υπάλληλο αριθμών 19. Στο Αλικάντι ήταν εκείνη η υπηρεσία. Βέβαια δεν είχα δικό μου γραφείο και έμεινα εκεί και υπηρέσαμε μέχρι το 2005 έκανα διάφορες δραστηριότητες ως νομικός, αλλά επίσης είχαμε πολλά να κάνουμε, να προετοιμάσουμε την υπηρεσία ε, πριν ξεκινήσει η υπηρεσία αρχιοθέτησης των ευρεσιτεχνιών και σημάτων μάλλον, των σημάτων. Κατόπιν πήγα στο γραφείο ευρεσιτεχνιών στο Μόναχο ε, ως επικεφαλής νομικής υπηρεσίας, είχα ζητήσει αυτή τη θέση διότι θεώρησα ότι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει την πνευματική ιδιοκτησία γενικά, εάν δεν ξέρει το δίκαιο των ευρεσταχνιών Τα σήματα, τα σχέδια στο Αλικάντε, αλλά έπρεπε κανείς να, πρέπει κανείς μάλλον να μάθει αυτά που είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας του μονάχου. Πέντε χρόνια λοιπόν ήμουν επικεφαλής της υπηρεσίας για όλα τα νομικά θέματα ε, όχι αυτά που έχουν σχέση με τις ευρυζηνίες καθηγητές, αλλά θέματα θεσμικά, θέματα εργασιακά κλπ. Οπότε, επανήλθα τώρα στην υπηρεσία αυτή της πνευματικής διαδικασίας το 11. Είχα συγκεκριμένες ε, αρμοδιότητες στην νομική υπηρεσία επομένως και συμβουλευτική υπηρεσία και Επίσης εργάστηκα και για το δεύτερο βάθμιο όργανο, γι' αυτό είμαι εδώ τώρα και από το 2015. Το 2015 ε, ασχολούμαι με αυτά τα θέματα με άλλους δύο συναδέλφους. Στις ε, πέντε γλώσσες εργασίας της υπηρεσίας έχουμε καταλήξει σε 600 αποφάσεις ως εισηγήτρια και Ω αναπληρώτρια εισηγήτρια, σύμβουλο σε άλλε 700. Δύο μεγάλες υποθέσεις έχω κρίνει. Πρώτα-πρώτα την ε, αίτηση για τα σήματα ε, σε σχέση με το Brexit για κάποια αναψυκτικά και επίσης άλλη μια απόφαση για την ομοιότητα βότκας νερού, υπόθεση iceberg. Αυτά όσον αφορά το τμήμα προσφυγών, όπου επίσης είχα μια ομάδα εργασία και ασχοληθήκαμε με την εναρμόνιση της διαδικασίας των προσφυγών. Και εγώ θέλω να προσφέρω σε αυτήν την υπηρεσία αυτά τα 25 χρόνια εμπειρίας ε, από σήματα και σχέδια και επίσης την εμπειρία από διαφορετικούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, την υπηρεσία μου στη πνευματική ιδιοκτησία, άλλο ευρωπαϊκό όργανο, επίσης ε, όσον αφορά τον ε, μηχανισμό σταθερότητας από το 2014 εκεί επίσης εργασμός ε, νομικός και κάποιες τις στατικές αλλαγές που σπούδασα ε, στην Οξφόρδη και εδώ και δύο εβδομάδες είμαι πιστοποιημένη μεσολαβητής. Δεν το βρείτε αυτό στο γραφείο γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Είμαι περήφανη για αυτό, είναι κάτι καινούριο, νέα προοπτική, δεν ορίζονται στη δουλειά μου και project manager. Θεωρώ ότι είμαι πολυδυναμική. Μάλιστα συνεργάζομαι με συναδέλφους από διαφορετικές ενωμές τάξεις, διαφορετικές χώρες. Αυτό κάτι γνώμη είναι μια ωραία πρόκληση. Μ' αρέσει η ομαδική προσπάθεια. Και ιδίω όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψει γιατί μόνο έτσι υπάρχει στεγανή απόφαση από πλευρά νομικής. Επίσης ε, μπορώ να δουλέψω υπό την χρονική πίεση των προθεσμιών, δεν φοβούν τεχνολογία και νομίζω ότι υπάρχουν ε, προκλήσεις για το πώς θα έχουμε τα μέσα εργασίας μας, ε, πώς θα τα βελτιώσουμε για να μπορούμε να, το έργο μας να διαδοθεί. Επίσης για να ολοκληρώσω να σου πω ποιο είναι το όραμά μου για αυτή τη θέση, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έγινε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και μάλλον γνωρίζετε ποιο είναι το στατικό πρόγραμμα ε, τον έρωτα του 25. Θέλουμε να είμαστε κόμβος ε, αριστείας και όσον αφορά το τμήμα προσφυγών θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους για την ποιότητα αλλά να έχουμε και συνέπεια θα πρέπει επίση να βοηθήσουμε με την ομολογία μας όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους πελάτες. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα κανάλια ε, επίλυσης διαφορών, γι' αυτό και πήγα για, στην υπηρεσία αυτή της διαμεσολάβησης. Ε, με ενδιαφέρει αυτό όσον αφορά την επίλυση των διαφορών στα πλαίσια της πνευματικής ιδιοκτησίας και έχω συνεργαστεί με διάφορους συναδέλφους άλλων χωρών για την πνευματική ιδιοκτησία με δικαστές και βέβαια ο καθένας σέβεται την αρμοδιότητα του άλλου αλλά επίσης και με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες που έχουν τμήματα προσφυγών και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πολύ ενδιαφέρουσα η προϋπηρεσία σας και η εμπειρία σας. Η κυρία Μέλχιορ ήταν η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που δεν έχουμε λόγο για το διορισμό σας, ε, να πούμε ναι ή όχι, η ομιλήτρια δεν μιλάει στο μικρόφωνο και δεν την ακούμε. Έχουν εκφραστεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Ας πούμε, η BMW, η Apple και κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονται. Υπάρχουν κάποιοι ε, που έχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμποδίζουν την καινοτομία και την πρόοδο της επιστήμης στην Ευρώπη ακριβώς γιατί επικαλούνται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Μιλήσατε για αριστεία, αλλά τι γίνεται με την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τι πιστεύετε για την αναλογικότητα και ναι, ναι, είναι σχετικό κριτήριο στην κατάθεση υποψηφιότητας για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Απάντηση. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είχα μια πενταετή εμπειρία στο Μόναχο, εξαιρετικά ε, χρήσιμη ε, έφυγα από τα σήματα και ε, τα σχέδια που ήταν το γνωστό μου έδαφος και πήγα ε, στις πατέντες, στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτές μπορεί να τα δει κανείς από διάφορες σκοπιές. Ορισμένοι θα πούν ότι είναι εργαλείο καινοτομία, διότι χωρίς την προστασία που φέρνει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορείς να είσαι πραγματικά βέβαιος για την επένδυσή σου όταν προσπαθείς να καινοτομήσεις, ιδιαίτερα όταν αυτό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Είναι ο μόνος τρόπος να εγγυηθείς ε, ότι θα έχεις κάποια ε, κέρδη από αυτό ε, το σύστημα. Βεβαίως, ορισμένοι επικρίνουν αυτό στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε ενιαίο δίπλωμα τεχνίας και αυτό το εργαλείο μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρυστεχνίας για να πετάξει έξω από ένα κλάδο τεχνολογικό τον ανταγωνιστή του και μόνο. Όλες οι προσπάθειες λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πάντα θα πρέπει να βρίσκεται σωστή ισορροπία. Βέβαια πάντα θα υπάρχουν πρόσωπα ή εταιρείε που θα καταχρώνται το σύστημα. Αυτό το βρίσκουμε και στα σήματα. Στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους έχουν μάλιστα ονομάσει patent trolls. Γιατί τρολάρουν. Για τα εμπορικά σήματα έχουμε καλύτερες δυνατότητες και από την νομοθεσία να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταχρήσεις του συστήματος. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει πάρει πολλά μέτρα για να ανοιχνεύονται ε, όλα αυτά σε κάποιους τομείς τεχνολογίας και να αντιμετωπίζονται. Στο δικό μας σύστημα, γιατί θέλουμε να είμαστε ε, κόμβος αριστείας για την πνευματική ιδιοκτησία, διότι είναι πάρα πολύ ε, ουσιαστική σημασία και για τις εταιρείες στην Ευρώπη, αλλά και όταν φεύγουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στο εξωτερικό. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο πλην άειλο και θα πρέπει να προστατεύεται πάρα πολύ σωστά με σχετικές ε, ένομες ε, παρεμβάσεις και μέσα και πραγματικά Βέβαια μετά από μια διετία είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι έχει λειτουργήσει πολύ καλά το νέο σύστημα. Πάντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα με τις ε, προκλήσεις ε, της ψηφιακής εποχής. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο και όλα αυτά τα ζητήματα που τίθενται από πλευράς επικράτειας τελευταία μας προσπάθεια, το τελευταίο εξάμεινο, ήταν να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο της τεχνολογίας, για να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα για να καινοτομούμε περισσότερο. Θα αλλάξουμε τελείως τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την ενημέρωση, για τις εταιρείες εκείνες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και χρειάζονται καλύτερη ε, καθοδήγηση. Νομίζω οι πολυεθνικές χρησιμοποιούν το σύστημά μας με πολύ καλό τρόπο και δεν χρειάζονται παραπάνω βοήθεια. Εμείς θα επικεντρωθούμε λοιπόν γι' αυτό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί εκεί είναι η πραγματική πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βος, Φως δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τις απαντήσεις που θα δώσετε στις ερωτήσεις μας. Χαίρομαι που συμμετέχετε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Έχετε όλη αυτή τη μακροχρόνια εμπειρία σε ε, αυτούς τους τομείς και κατά την άποψή μου θα είχε νόημα να μάθουμε την άποψή σας για το μέλλον. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε εμείς ή εσείς που τα αναφέρατε για να είμαστε πιο έτοιμοι και ποιες είναι οι πιο επίγουσες αλλαγές τις οποίες θα πρέπει να προβούμε για να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέλλον. Δεν θα πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια θέματα του παρελθόντος και απλώς να τα βελτιώνουμε. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, χρειαζόμαστε νέες δομές. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Διότι όπως είπα, η μεταρρύθμιση είναι μόλις ηλικίας δύο ετών. περιλαμβάνει πολλές ε, ρηξικέλευτες αλλαγές. Για παράδειγμα, όταν αποφασίσατε να καταργηθεί η απέτηση γραφικής αναπαράστασης ενός σήματο, άνοιξε ένα τεράστιο τοπίο πολυμέσων, βίντεο, μουσικής ε, που μπορούν να αρχιοθετηθούν και ένας τελείως νέος τρόπος ε, σκέψης. Αλλά αυτό είναι το μέλλον. Το μέλλον, το μέλλον είναι αυτό που βλέπετε στο YouTube, ένα τραγουδάκι που ε, ακούτε όταν μπαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ. Ίσως το μέλλον να είναι και η μυρωδιά, εάν το επιτρέψει η τεχνολογία, και η γεύση. Οπότε ε, ανοίξατε ένα τελείως νέο πεδίο. Φανταστείτε εμάς που για 25 χρόνια ζητούσαμε κάτι το οποίο μπορούσες να αγγίξεις, κάτι απτό ως γραφική αναπαράσταση. Είναι μία επανάσταση πραγματική. Ε, προβλέπει το κατά κάποιο τρόπο το πώς είναι η επιχειρήση τώρα και πώς θα είναι στο μέλλον ε, όλη αυτή η νέα τεχνολογία που θα εμφανιστεί Κατά μία είναι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αντιδράμε όσον αφορά αυτά τα σήματα με ικανοποιεί γιατί ούτε τα έχουμε περιορίσει, ε, υπάρχουν αρκετά που έχουν ε, καταχωριστεί και αυτό είναι καλό για το μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοράμε παροπίδε ε, μπροστά σε όλες αυτές τις νέες δυνατότητες. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Όπως υπόθηκε και στην προηγούμενη ερώτηση, ούτω ώστε να έχουμε υπόψη μας τις ε, απόπειρες ε, κατάχρησης του συστήματος. Σε αυτό το πεδίο δεν είμαστε απόλυτα ε, έτοιμοι για αυτό το πιο ευρύ ανταγωνισμό, αντί να χρησιμοποιήσω τη λέξη τρόλ, ευρύ ανταγωνισμό. Θα μπορούσαμε να... Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά την φήμη και τα γνωστά εμπορικά σήματα. Η φήμη ε, χτίζεται με χρόνια επενδύσεων, διαφήμισης, ε, δέσμευσης, επιμονής ε, κτλ. Οπότε δικαίως πρέπει το νομικό μας σύστημα να τα προστατεύει, αλλά ίσως να μην τα προστατεύουμε αρκετά. παρέχονται μετά από εκατοντάδες αποδεικτικά στοιχεία και φυσικά τα επαναλαμβανόμενα σήματα Διάφοροι προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν ε, χάρη στην ε, καλή τους φήμη. Ίσως να υπάρχουν και άλλα συστήματα στον κόσμο που θα μπορούσαμε να συμβουλευτούμε. Μήπως υπάρχει κάποιο τρόπος να φτιάξουμε κάποιο λίστα ή κάποιο δυναμικό μητρό ε, γνωστών σημάτων ούτως ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην χρειάζεται κάθε φορά να προσκομίζουν όλα τα στοιχεία για να μας πείσουν. Το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο έχει βρει έναν ωραίο τρόπο. Λέει ότι αν έχει ήδη εκτιμηθεί, αξιολογηθεί ε, ότι υπάρχει κάποια φήμη, μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτήν. Ήδη πριν από 10 χρόνια. Αυτό ήδη είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να προστατεύσουμε καλύτερα τα σήματά μας. Και τέλος έχω να πω ε, ότι οι προσπάθειές μας είναι κυρίως ε, στοχευμένες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια Χρειάζονται παροχή γνώσεων, χρειάζονται να τους δώσουμε παραδείγματα, να τις καθοδηγήσουμε, γιατί εκεί θα γεννηθούν οι μελλοντικές δουλειές στην Ευρώπη, ειδικότερα οι καινοτόμε ε, μικρές επιχειρήσεις, που ίσως καινοτομούν ε, σε επίπεδο ποιότητας και δεν επιλέγουν ε, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καταστρεπτικό, να καταστρέψει μια startup μόλις αυτή ξεκινάει να υπάρχει πέρυσι βρέθηκα στην Κύπρο για μια διάσκεψη σε σχέση με τις μικρές γεωργικές επιχειρήσεις που επενδύουν σε ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή προϊόντα με γεωγραφική προέλευση, με ονομασία προέλευση, συγγνώμη ήταν περίεργο. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τι, πώς προστατεύονται με ένα σήμα, πώς προστατεύονται ως γεωγραφική ένδειξη, τι σημαίνουν όλα αυτά, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και ακόμη και μετά τη διάσκεψη συνεχίσαμε να συζητάμε, διότι δεν ήταν αρκετοί για να καταλάβουν και υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να καταλάβουν αυτές οι εταιρείε και αυτό αποτελεί τεράστια, αυτή η γνώση αποτελεί τεράστια επένδυση για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βόλκεν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Και ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Έχετε τεράστια εμπειρία. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχω μια γενική και μια πιο ειδική ερώτηση. Η πιο γενική μου ερώτηση είναι τι προβλήματα διακρίνετε, θεωρείτε ότι θα υπάρξουν στο μέλλον στον κλάδο σας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα συναντήσουμε στο μέλλον και πώς ε, εμείς πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και η πιο η δική μου ερώτηση Ένα από τα προβλήματα είναι ότι πρέπει να προσαρμόσουμε το κλασικό μας σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας ε, στην ταχύως μεταβαλλόμενη οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο σε δεδομένα. Ποια είναι η αποψή σα, τι πρέπει να κάνουμε, τι είναι αναγκαίο να κάνουμε και είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το σύστημα εμπορικών σημάτων και σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετωπίζει ως μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα τις ποσότητες, τον όγκο το γραφείο είναι μια ιστορία επιτυχίας. Πέρυσι είχαμε την 25η επέτειο του γραφείου μας και θυμάμαι ότι το, τον πρώτο μήνα προβλεπόταν ότι θα λάμβανε 15.000 αιτήσει ε, το γραφείο και αυτό το θεωρούσαν θετικό σενάριο και σε τρεις μήνες είχαμε 45.000 δεν ξέραμε πού να βάλουμε όλα τα αρχαία τότε δεν είχαμε ακόμα την τεχνολογία με τους υπολογιστέ που έχουμε σήμερα. Πέρυσι δεχθήκαμε πάνω από 160.000 αιτήσει. Οι προκλήσεις, που, οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αν δείτε την ε, ονομασία, την χώρα προέλευση. και πώ εξελίσσεται αυτό, οι Ευρωπαίοι υπάρχουν όσο υπήρχαν και παλιότερα. Όταν ξεκινήσαμε το γραφείο το 1996 και αρχίσαμε να λαμβάνουμε αιτήσει, η Κίνα ήταν νομίζω στην εκατοστή δέκατη θέση και σήμερα είναι στην τρίτη. Και αυτό δημιουργεί διάφορες δυσκολίες, αλλά η ποσότητα νομίζω ε, ότι είναι ε, ε, το πιο δύσκολο. 19.000 ενστάσεις, 3.000 ακυρώσεις, 3.000 εφέσεις και είμαστε μόλις 19 ε, αυτοί που λαμβάνουμε αποφάσεις. Φυσικά σε 23 επίσημες γλώσσες. Δηλαδή οι ποσότητες, ο όγκος που πρέπει να διεκπαιρεώσει το σύστημά μας. Το σύστημά μας ε, έχει να αντιμετωπίσει και όλες τις ε, ε, διαφορές νοοτροπίας με τις αιτήσεις που έρχονται από την Ασία, από την Νότιο Κορέα, σχέδια που έρχονται από την Νότια Κορέα, από την Ιαπωνία. Δεν έχουμε τέτοια συστήματα εναρμόνισης. Το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, νομίζω ναι. Έχουμε συμπεριλάβει στο στρατηγικό μας σχέδιο διάφορες προτάσεις και πρωτοβουλίες κλειδιά που θα μας βοηθήσουν ειδικότερα σε τεχνολογικά θέματα. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι όταν εμείς νομοθετούμε σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, το πράττουμε με γνώμονα την επικράτεια. Πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία της online χρήσης του σήματος, των online επιθέσεων, των online παραβιάσεων, της online κυκλοφορίας απλαστών προϊόντων που εκμεταλλεύονται βασίζονται στην ε, φήμη ενός ε, καθιερωμένου εμπορικού σήματος. Και εκεί έγκυται το η πραγματική δυσκολία. Οπότε πρέπει να εξελίξουμε περισσότερο τα εργαλεία ε, επιβολής και άλλες πρωτοβουλίες που μας προσφέρει η ψηφιακή οικονομία. Φυσικά, ο νόμος δεν είναι πανάκια. Εμείς στο τμήμα προσφυγών λαμβάνουμε δευτεροβάθμιες αποφάσεις και εμείς μαζί με το δικαστήριο και το οποίο επίσης μπορεί να προσβάλλει τις δικές μας αποφάσεις πρέπει να έχουμε γνώση του ότι πρέπει να δείξουμε δημιουργικότητα. Για παράδειγμα, αν ένα εμπορικό σήμα πρέπει να αποδείξει ότι έχει χρησιμοποιηθεί και έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιβάλλον online πρέπει να δείξεις και εσύ ότι είσαι πιο ανοιχτό Δεν μπορείς να απαιτήσει ε, να έχει απόδειξη για τη χρήση μόνο σε, ε, στον έξω κόσμο. Αλλά είμαι αισιόδοξη. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι άλλο. Ο κύριος Βόσου. Μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο της προσοχής μας. Τι ακριβώς εννοείτε, ότι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τους παρέχουμε ε, κάποια υπηρεσία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις ενημερώνουμε καλύτερα, να τις ε, βοηθάμε περισσότερο Τι να κάνουμε δηλαδή όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Το νέο μας στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει ειδικό πυλώνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά βασιζόμαστε και στην πρωτοβουλία της Κομισιόν που θέλει να θέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής. Όταν δει κανεί του ετούντε για σχέδια ή για εμπορικά σήματα, ε, πρόκειται για μεγάλε εταιρείε. Ξέρουμε ότι το σύστημα ευαισθητοποίησή μα, το σύστημα ενημέρωση μέσω τη ιστοσελίδα, λειτουργεί μια χαρά. Αλλά τι συμβαίνει όταν ένα μικρός Έλληνας παραγωγός ενός εξαιρετικού ελαιόλαδου αποφασίζει ε, μια μάρκα που ήδη χρησιμοποιείται και ε, ε, τον προσβάλλει κάποιος ε, αντίπαλος ε, και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει αν μπορεί να απαντήσει στα ελληνικά και Εκεί παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων και όταν μπαίνουν στο σύστημα δεν έχουν γνώση. Οπότε σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο παρατηρούμε διάφορα ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε, ευαισθητοποίηση όπως είπατε, ε, εκπαίδευση, ε, αρρωγή. Φυσικά δεν παρέχουμε νομική ε, στήριξη, δεν είναι αυτός ο στόχος ύπαρξής μας, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με τους απλούς ανθρώπους, αυτούς που εργάζονται στα εθνικά γραφεία, στα κράτη-μέλη μας, οι οποίοι γνωρίζουν τις καταστάσεις, ήδη εργάζονται με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να κάνουμε έναν ε, βρούμε μια κοινή γλώσσα όταν συζητάμε για τις διάφορες υποθέσεις. Ε, να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ίσως να μην χρειάζεται τελικά ένα ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα, ίσως να πουλάνε τα προϊόντα τους σε ένα-δυο κράτη-μέλη, ίσως να μην χρειάζονται ευρωπαϊκό σήμα. Ίσως να μην είναι απαραίτητο για, για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε ε, πρέπει να βρεθεί μία γλώσσα προσαρμοσμένη. Αυτό πιστεύω είναι η βασική γραμμή της στρατηγικής μας. Τώρα μου λέτε γιατί το τμήμα προσφυγών ε, ασχολείται με κάτι τέτοιο. Διότι όταν ξεκινάει ε, η διαμαχνίας υπόθεσης υπάρχει πολύ φόβος. Πόσο θα κοστίσει, χρειάζομαι δικηγόρο και ο δικηγόρος πρέπει να μιλάει τη γλώσσα ε, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, πώς θα το πληρώσω. Οπότε τα παρατάω και ξαφνικά τα δικαιώματα τα ε, βουτάει κάποιο άλλος. Ε, γιατί, διότι φοβούνται να πάνε δικαστικά. Γι' αυτό έχουμε εισάγει την εναλλακτική επίλυση διαφορών που είναι φθηνή, απόρριτη, πολύ γρήγορη. Έχουμε διαμεσολαβητές που μιλάνε όλες τις γλώσσες, με πολύ, που είναι πολύ έμπειροι έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να πάνε δικαστικά για κάτι και ε, έτσι βοηθάμε ε, και ε, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και έτσι έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση εναλλακτική επίλυση διαφόρων. Θα μπορούσα να σα πω και άλλα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο, για τι απαντήσει σα που ήρθατε να μα δείτε. Ήταν χαρά μα που σα είδαμε και καλή επιτυχία στην επόμενη φάση. Μέλγκαρτ, εγώ σας ευχαριστώ και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για πολύ περισσότερη ώρα για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέσμα σας διάταξη. Ε, με μεγάλη μας χαρά ε, καλώς όρισε εδώ η Μαργαρίτα Βεστάκερ για να μας μιλήσει. Κάπως έτσι δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Βέστεγερ, και μεγάλη μας χαρά έχουμε αυτή την ευκαιρία για αυτή την ε, νωρίς νωρίς ανταλλαγή απόψεων και, και προσωπικά χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας ε, ακούσω σε αυτή μας την τελευταία εβδομάδα. Που έχουμε. Οπότε, η ψηφιακή εποχή. Το και πώ θα προσαρμοστούμε, αυτό είναι κάτι που αφορά εμά όλου του ε, νομοθέτε. Και όπω ξέρετε, έχουμε αρχίσει τώρα να συντάσσουμε κάποιε εκθέσει για την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε και εμεί να βάλουμε λιθαράκι για αυτή την υπόθεση. Οπότε να σα δώσουμε τώρα το λόγο για την εισηγησή σα και κατόπιν να ακούσουμε τι ερωτήσει των συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Και μετά θα έρθει η ώρα των ερωτήσεων θα έχουμε ερώτηση και απάντηση μία-μία. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, δηλαδή τίποτα είναι συναισθηματικά φορτισμένη η εβδομάδα αυτή. Αλλά, ευχαριστώ που με καλέσατε. Πολύ σωστή ώρα που με καλέσατε. Όπως ξέρετε έχουμε 19 Φεβρουαρίου, οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει την λευκή βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σχετική στρατηγική δεδομένων. Οπότε πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις σας και να ακούσω τι έχετε να προτείνετε πριν γίνει η έγκριση και της Λευκής Βίβλου αλλά και της σχετικής στρατηγικής. Τώρα, για την τεχνητή νομοσύνη προσέχουμε δύο τινά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε το στόχο της ευκαιρίας, τι βοηθάει την κοινωνία, την ε, υγεία, την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, για την μόλυνση της ε, πόλης και πάρα πολλά άλλα θέματα που μας βοηθά σε αυτά. Είναι η τεχνητή νομοσύνη, γιατί είναι τόσα πολλά δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούμε, που θα ήταν αδύνατο σε ατομική βάση κάποιο να τα επεξεργαστεί. Επομένω, τώρα μπορούμε να έχουμε καλύτερη αναγνώριση των τεχνιών, μπορούμε να ζυγίσουμε τι δυνατότητε που υπάρχουν. Επομένω, πολλά, πολλά θα προκύψουν θετικά. Οπότε, οι δύο προσεγγίσει που έχουμε είναι το οικοσύστημα εμπιστοσύνη και οικοσύστημα αριστεία. Για το πρώτο. Εμπιστοσύνη. Έτσι θα καθισχαστεί ο πολίτης ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει και χρησιμοποιείται έτσι που να σέβεται τα δικαιώματα και τις αξίες. Αμφιγεδία κρίσεων, προστασία ιδιωτικού βίου, ασφάλεια και αξιοπιστία. Πολύ σημαντικό γιατί η εμπιστοσύνη προς την τεχνολογία κάθε μέρα και μειώνεται. Έχουμε ένα σωρό πηγέ από τι οποίε προκύπτει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμο ότι τα πιο σημαντικά είναι στεγανά. Και μετά έχουμε το θέμα της αριστείας, τι ευρωπαϊκές δυνατότητες, ούτως ώστε να φτιάξουμε όπω θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη και από πλευρά ανταγωνιστικότητα, ούτω ώστε να μπορούμε να καθιερώσουμε κάποια πρότυπα διεθνώ, γιατί αν το κάνουμε αυτό το θα τα καταφέρουμε. Αλλιώς δεν θα έχουμε την ε, γνώση, τις δυνατότητες, τις δεξιότητες να τα καταφέρουμε. Οπότε τι προϋποτίθεται ούτω ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την εξέλιξη ε, και την πρόοδο της τεχνητής στην Ευρώπη. Θέλουμε δεδομένα ποιοτικά για την ε, πριν την νοημοσύνη θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα των επενδύσεων στην έρευνα. Σήμερα δεν μπορούμε να κοντράρουμε τη ΣΥΠΑ όσον αφορά τις ε, επενδύσεις στην έρευνα. Να στοχεύουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά την έρευνα, όσον αφορά την καινοτομία, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες στην Ευρώπη. Αλλιώς, αν δεν τα καταφέρουμε, τότε χάνεται μεγάλη ευκαιρία. βγούμε χαμένοι. Επίσης, θα πρέπει κατά να κάνουμε και για τον ε, δημόσιο τομέα. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι ο σεβασμός των αξιών, η διακρίσεων δηλαδή είναι κάτι που ισχύει καθημερινά στην πράξη. Διαφάνεια, υπευθυνότητα και επίσης με αυτές τις δεξιότητες θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, εκπαίδευση τι ε, τις και στα ψηφιακά και όχι μόνο για τους προχωρημένους ε, μηχανικούς ας πούμε αλλά και για όλο τον κόσμο να μπορεί όλος ο κόσμος να καταλάβει με τι έχουμε να κάνουμε. Επίση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο χρειάζεται ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η εμπιστοσύνη, γιατί αυτοί που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη ήδη υπόκεινται στο γενετικό δίκαιο. Και για την προστασία των δεδομένων, για την προστασία του βίου, για τις διακρίσεις, ισότητα των ε, ναι των δύο φύλων, ε, την ερμηνεία των κανόνων, για όλα τα προϊόντα που σχέση την νοημοσύνη. Όλα αυτά θα καλυφθούν από την νομοθεσία που σας είπα. Το θέμα είναι ότι είναι τέτοια η φύση της νοημοσύνης που γίνεται πιο δύσκολο να υλοποιηθούν όλα αυτά να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχουν αυτά τα χαριστικά black box Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιο μπορεί να επικαλεστεί ένα δικαιωμά δεν ξέρει εναντίον ποιου θα προσφύγει, για να αυτό καταπατηθεί. Άρα χρειάζεται να υπάρξει σωστή νομοθεσία που να καλύπτει τους σχετικούς ε, κινδύνου και όπου υπάρχει παραθυράκι να το διορθώσουμε. Και ενώ τέλο πάντων. Οπότε μπορεί επίση να ισχύει ότι υπάρχουν ακριβώ και αυτά τα κενά, κάποια θέματα λέτε δηλαδή που δεν καλύπτονται. Αυτά θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε δεν υπάρχει πραγματικά εσωτερική αγορά. Άλλο. Πού θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Γιατί ίσως ε, έχω μόνο jazz δεκαετία του 50 από το ίντερνετ. Δεν μπορώ να βρω δηλαδή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα ε, ένα soundtrack ε, τη Eurovision. Αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα εάν είναι ζήτημα μιας εφαρμογής ζωή σε θανάτου. Αν, αν ε, κάτι δηλαδή το οποίο είναι κακόηθες, ε, ε, αυτό είναι διαφορετικό και εκεί πέρα είναι πολύ πιο μεγάλη από το θέμα της μουσικής που ανέφερε στην αρχή. Βέβαια, από αυτά τα παραδείγματα διαπιστώνεται ότι θα πρέπει κανείς να δει τι ισχύει. Πότε υπάρχει ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος ο μεγάλος, ο μεσαίος, ο μικρός ή καθόλου κίνδυνος. Αυτά θα πρέπει να συζητηθούν επίσης. Να δούμε τι γίνεται με τον δημόσιο τομέα, τις ε, υπηρεσίες, ε, δημοσιο ενδιαφέροντος, κάποιες υπηρεσίες, Αντίστοιχε κατά πόσο είναι στα στάνταρ που πρέπει, τα υψηλά όσον αφορά τη διαφάνεια, ή την ε, υποχρέωση λογοδοσία. Ίσως εκεί δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά επειδή είναι το δημόσιο και επειδή είναι ο δημόσιος Κορβανά θα πρέπει εκεί να είναι υψηλά τα πρότυπα. Επίσης, θα είναι αναγκαίο να εξετάσουμε καλύτερα κάποιες ε, τεχνολογίες ιδιαίτερα δύσκολες όπως την αναγνώριση του προσώπου. Εκεί υπάρχει και προβληματισμός μεγάλος. Είναι θέμα προστασίας δεδομένων και αξιών όπως το δικαίωμα του συναθρίζεστε. Εδώ αλλάζει η προσέγγιση για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε και ο κόσμος να καθυσυχαστεί ότι με τη σωστή χρήση δικαιολογείται αυτό που θα γίνεται Τώρα όσον αφορά την αξιοπιστία και την ασφάλεια θα έχουμε στη Λευκή Βίβλο μια σχετική έκθεση για αυτό, για αυτό το πλαίσιο αξιοπιστίας και ασφάλειας. Ήδη ξεκινήσαμε την μελέτη επιπτώσεων για να ζηγήσουμε το κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Και για ασφάλεια και για αξιοπιστία. Ίσως τα κλείσουν όλα αυτά με κάποιον σχετικό κανονισμό για το δημόσιο, για τον κίνδυνο κλπ. Οπότε και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, ανιχνευσιμότητα των δεδομένων, την ποιότητά τους, να δούμε ακριβώς με τι δεδομένα θα πηγαίνουν, θα δημιουργούνται οι αλγόριθμοι, μήπως κάτι λείπει, γιατί πολλές φορές κανείς προβληματίζεται με την ποιότητα των δεδομένων γιατί ίσως τα δεδομένα που δεν έχει κανείς αυτά είναι που δημιουργούν το πρόβλημα γιατί έτσι τα πράγματα γίνονται λιγότερο αντικειμενικά. Επίσης διαφάνεια όσον αφορά την, τις ικανότητες ή τα όρια των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοια όρια και περιορισμοί. Επίσης διαφάνεια σε σχέση με τον πολίτη που την χρησιμοποιεί την ε, τεχνητή νομοσύνη ή επηρεάζεται από αυτή να υπάρχει σχετική εποπτεία. Μιλά κανεί με ρομπότ, μιλά κανεί με ε, φυσικό πρόσωπο. Α, τις προάλλε μου συνέβη αυτός με κάποια υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών. Δεν ήταν ε, προφανές, δεν, δεν μπορούσα να καταλάβω αν μίλαγα με άνθρωπο. Χαζό αυτό. Και τελευταίο αλλά σημαντικό όσον αφορά τις προτεραιότητες και τις καταπροαπαιτούμενα είναι το τι θα πρέπει να εφαρμοστεί, να ισχύσει νομοθετικά γιατί όπως σας είπα βέβαια να ακούσω την απόψή σας είπαμε ότι καλύτερα να έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά να τις εφαρμόσουμε παρά να έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο από σημεία που θέλουμε να εφαρμοστούν αλλά δεν γίνεται να τα εφαρμόσουμε. Α, δύο λόγια τώρα όσον αφορά τη στατική για δεδομένα και για το νομοθέτημα για τι ψηφιακέ υπηρεσίε η στατηγική πηγάζει από το ότι οι ψηφιακέ τεχνολογίε και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν σχέση, βασίζονται σε δεδομένα πολλέ φορέ σε τεράστια ποσότητα δεδομένων, οπότε θα πρέπει αυτά να διατίθενται στην Ένωση σε διάφορου τομεί, ή κλάδου, και για αυτό επεξεργαζόμαστε αυτή τη στρατηγική για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση, χρήση, αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στην Ευρώπη. Και εν προκειμένου να σιγουρέψουμε ότι η καινοτομία εδώ για τα δεδομένα ωφελεί, ε, καλύπτει τους κοινωνικού μας ε, στόχους και να εξασφαλίσουμε ότι και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων. Και είπαμε στις 19 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσουμε και αυτή τη στρατηγική για τα δεδομένα. Οπότε αυτό πάει και στην καινοτομία και στο θέμα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Να οργανώσουμε τη χρήση, την πρόσβαση στα δεδομένα. Αυτό θα καθορίσει τις δυνατότητές μας για καινοτομία στο μέλλον. Επίσης, πολλές φορές η συγκέντρωση των δεδομένων και η μεταβίβασή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι μπορεί κάποια επιχείρηση να ορθώσει ανάστημα εναντί κάποιου γίγαντα της αγοράς και θα πρέπει μας όλα αυτά να γίνουν με τον σωστό τρόπο για να δώσουμε δυνατότητε ανταγωνισμού σε τέτοιου είδου αγορά που κυβερνάται από τα δεδομένα. Για υποδομές, είπαμε υπάρχει και μια τέτοια διάσταση. Η ψηφιακή οικονομία είναι δεδομένη. Αλλά πρέπει να αυξηθούν και οι δυνατότητες. Blockchain, το ίντερνετ των πραγμάτων, όλα αυτά να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις. Σχέσεις με τρίτες χώρες. Να δούμε τι θα γίνει με την κατάργηση των πολιτικών εντοπισμού των δεδομένων. Να δούμε τι θα γίνει με τους κανόνες που έχουμε για τα δεδομένα, τα στάνταρ, προστασία δεδομένων, ασφάλεια αυτών. Α, και κάτι άλλο. Για αυτό το τελευταίο το νομοθέτημα, δηλαδή για τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες. Ο σκοπός είναι να προσαρμοστούμε. Γιατί αλλάζει το τοπίο όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες και να υπάρχει ε, ασφαλεία δικαίου, εναρμόνιση περισσότερη. Να προστατεύσουμε δηλαδή τον Ευρωπαίο και να είναι πιο ολοκληρωμένη η εφαρμογή του νόμου. Πολλά θέματα που έχουμε δική μας πρωτοβουλία να τα ξεκινήσουμε και θα πρέπει να είμαστε στοχευμένοι σε αυτή την προσπάθεια γιατί έχουμε αυτό το γενικό νομοθέτημα για τα ψηφιακά και να δούμε τι θα καλυφθεί ποιος μπορεί να καλυφθεί, ποιος θέλει να καλυφθεί. Οπότε περιμένω ανυπόμονα και τις ερωτήσεις σας, αλλά και τις προτάσεις σας. Γιατί τώρα είναι η σωστή στιγμή να μπορούμε να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές στην προσπαθία μας. Thank you very much indeed for an excellent... Εγώ σας ευχαριστώ. Εξαιρετική η παρουσίασή σας και έχω και μακρύ κατάλογο ερωτήσεων. Ε, προσωπικά, έχω και μακρύ κατάλογο μιλητών που θέλω να κάνω ερωτήσει. Ο κύριος Ράντεφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Ε, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, φυσικά χρόνια πολλά και καλή επιτυχία στη θητεία σας. Ε, уважаема госпожо комисар, Αξιότιμη ε, κυρία Επίτροπε, επαναλαμβάνω, σας εύχομαι ε, καλή θητεία και καλή χρονιά. Έχουμε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόεδρος Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είπε ότι η νέα νομοθεσία θα βασιστεί στα όσα έχουν ήδη γίνει ως προεργασία για τα ψηφιακά προϊόντα και τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά. Η πρόταση αυτή είναι φωτοτυπία της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και πότε πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει περαιτέρω εναρμόνιση ή προτάσεις τουλάχιστον για τις ψηφιακές συμβάσεις και ποια θα είναι η νέα νομοθετική προσέγγιση απέναντι στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα την τεχνολογία blockchain. Και πώς θα ενημερώνονται οι πολίτες, πάντα θα πρέπει να ενημερώνονται από τον πάροχο των υπηρεσιών, ε, έτσι ώστε να ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτές. Τι αλλαγές θα φέρετε, γιατί ακόμα γινόμαστε μάρτυρες καταστάσεων όπου οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν απολύτως ε, τι ισχύει και τι ε, υπάρχει σχετικά με μια σύμβαση που υπογράφουν, προβαίνουν σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Και υπάρχει και ένα της περιορισμένης ευθύνης αυτή θα παραμείνει ή στη νέα ε, πρόταση θα επιζητείτε περισσότερη εναρμόνιση. Ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις σας. Ευχαριστώ. On, ε, Απάντηση για την νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ρωτάτε. Αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, είναι καθοδόν. Όπως γνωρίζετε από τις ε, επιστολές που μας έστειλε η Πρόεδρος ε, για την ανάθεση της εντολής μας. Έχουμε πυροθεσμία 100 ημερών για να κάνουμε τις προτάσεις μας. Αυτό ε, τονίζει και την ανάγκη να υπάρξει μια ολόκληρη στρατηγική για τα δεδομένα. Και εκεί εστιάζουμε τώρα. Δεν έχω να σας δώσω οριστικές ε, απαντήσεις σε καμία περίπτωση, αλλά θα το δείτε αυτό από το νομοθέτημα. Έχετε δίκιο να λέτε ότι πολλοί καταναλωτές αισθάνονται ότι έχουν δικαιώματα τα οποία αγνοούν και ακόμα περισσότερο αγνοούν πώς θα τα επιβάλλουν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενημερωθούν για το τι περιλαμβάνεται στους όρους και οι προϋποθέσεις που εκ των προτέρων έχουν υπογράψει. Δεν έχει ολοκληρωθεί, σας είπα, αυτή η προσπάθεια. Τρέχει. Το δεύτερο, ε, ποια είναι η επίπτωση του γεγονότος ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν αλλάξει ε, ραγδαία την τελευταία 20 ετία. Μπορεί να χρειάζεται ενημέρωση η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, πάντω δεν έχουμε λάβει ακόμα σχετική απόφαση. Σημειώνω τη φιλοδοξία τη δική σα Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για ε, να εκπονήσετε από κοινού μαζί μα ε, την νομοθεσία για τι ψυχιακέ υπηρεσίε. Εμεί δεν θέλουμε να έχουμε πολύ αυστηρού ή άκαμπτου στόχου από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φεστάγκερ για την παρουσίασή σας ε, για αυτό το συναρπαστικό θέμα και πιστεύω μας περιμένουν συναρπαστικές εποχές μαζί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα διότι η τεχνητή νοημοσύνη και η σχετική διαχείριση και η χρήση της, πώς θα χρησιμοποιήσουμε και θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα δεδομένα θα είναι καθοριστικά και για την δυνατότητα που θα έχουμε να καινοτομήσουμε και να ανταγωνιστούμε και παγκοσμίω. Και της, ε, και να αξιοποιήσουμε την ε, δική μας εσωτερική αγορά και τη διεθνή αγορά. Εμένα με ενδιαφέρει η ευθύνη της ασφάλειας των προϊόντων. Ειδικότερα ε, το σήμα που απαιτείται για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις, πώς θα έχουμε εναρμόνιση ε, πώς θα εξοπλιστούμε νομικά ούτως ώστε σε αυτό τον κλάδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να ε, ε, αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ε, και να κάνουν τους σχετικούς ελέγχους. Επίσης το data pool που χρειαζόμαστε να μοιραστούμε δεδομένα επίσης. Ξέρουμε ότι το μόνο 20% των δεδομένων χρησιμοποιούνται, διότι μόνο αυτά είναι διαθέσιμα. Πώς θα οργανώσει κανείς ένα τέτοιο pooling and sharing δεδομένων, μια συγκέντρωση και διαμοιρασμό δεδομένων και τέλος ε, η ανάπτυξη του ΓΕΑΕΚΣ δεν θα μπορούσε και αυτό να εξυπηρετήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους και να τα διαθέτουν με ασφάλεια. Οπότε αυτή είναι η ερώτησή μου σε αυτή τη στρατηγική για την τεχνική νοημοσύνη. Πώς θα διασφαλίσουμε την λογοδοσία, την ευθύνη και την ασφάλεια των δεδομένων. Ευχαριστώ. first and foremost, I very much... Λοιπόν, πρώτον, συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Μόνο όταν ε, είναι επικίνδυνα κάποια προϊόντα ότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή να παραβιάσουν θεμελιώδεις αξίες, μόνο εκεί υπάρχει νομοθετικό ε, πλαίσιο αυστηρό, οπότε πρέπει να υπάρχει κάποια αναλογικότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία να εξετάζουμε τα πιθανά, να βρούμε τα πιθανά ε, ρυθμιστικά και κανονιστικά κενά, διότι ήδη πολλά προϊόντα σήμερα καλύπτονται από τον κανονισμό που έχουμε ήδη. Το δύσκολο όμω είναι ότι η διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ενός προϊόντος είναι αυτή που του δημιουργεί πρόβλημα. Ε, ως προς αυτή είναι πιο δύσκολο να ασκήσει κανείς δικαιώματα. Είναι πιο δύσκολο να ασκήσει κανείς ε, ε δικαιώματα όταν μιλάμε για μια τεχνολογία εκμάθησης, για παράδειγμα, ή που εξελίσσεται. Ε, υπάρχει νομοθεσία που καλύπτει του σκοπού, αλλά χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τι κενά έχουμε όταν ε, εξελίσσεται μια κατάσταση, όταν αλλάζουν τα πράγματα και ξαφνικά ο κανονισμό μα δεν ε, προσαρμόζεται στην τρέχουσα κατάσταση. Αυτό κάνουμε τώρα. Τώρα για το ζήτημα των δεδομένων, λέτε πολύ σωστά ότι ήδη τώρα έχουμε πολλά δεδομένα διαθέσιμα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Πολλές επιχειρήσεις ε, έχουν αυτή την αίσθηση ότι κάθονται πάνω σε μια φλέβα χρυσού αλλά δεν ξέρουν πώς να την αξιοποιήσουν. Οπότε τελικά δεν είναι χρυσό, είναι τίποτα, διότι δεδομένα που δεν μένουν να χρησιμοποιείται δεν έχουν καμία αξία. Οπότε μέρος αυτού είναι να μπορείς φυσικά ως μικρή επιχείρηση να πεις τι θα κάνω, πώς θα το κάνω όλο αυτό, πώς θα τραβήξω τα δεδομένα να τα αξιοποιήσω. Για παράδειγμα, αν ε, έχεις ένα μεγάλο ε, αλυσίδα λιανικής πώλησης και μικρά μικρούς ε, λιανοπολιτές. Η μεγάλη αλυσίδα έχει πολλές δυνατότητες, πολλά δεδομένα και δυνατότητες να τα, να τα εκπεξεργαστεί. Οπότε είναι πολύ ισχυρός ανταγωνιστής ενώπιον των καταναλωτών. Αν μικρότεροι μπορούσαν να έχουν τέτοια δεδομένα θα μπορούσαν να γνωρίζουν και να καταλάβουν καλύτερα την αγορά και τους πελάτες. Και έτσι να είναι ισχυρότεροι ανταγωνιστές προς τη μεγάλη επιχείρηση. Ε, οπότε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα. Δεν είναι νομικά ακριβώς ε, τα εμπόδια, αλλά ε, περισσότερο μια ιδέα είναι τα εμπόδια αυτά, θεωρητικά. Στην ανθρώπινη δηλαδή υποδομή χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά, όχι στη φυσική υποδομή με μια εξαίρεση. Ένα τα συναρπαστικά πράγματα όσον αφορά το είναι η πρόσβαση στους μικρότερους παρόχους υπηρεσιών στην Ευρώπη ούτω ώστε εκεί να εφαρμοστούν κάποια μέτρα τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ε, αντιληφθούν ότι υπάρχουν και ε, εναλλακτικές όσον αφορά τους ε, μεγαλύτερους παρόχους υπολογιστικού νέφους, δηλαδή cloud, υπηρεσιών cloud, ότι να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι υπάρχουν και μικρότεροι παρόχοι cloud που προσφέρουν πρόσβαση στα δεδομένα και κρυπτογραφημένα. Το βασικό δηλαδή είναι ο κόσμος να καταλάβει πώς μπορεί να διαμοιραστεί και να αντλήσει δεδομένα και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα. Ειδικότερα και δεδομένων των αλλαγών που θα επέλθουν πιθανότητα μέσα στην επόμενη πενταετία ή δεκαετία. Δηλαδή θα αποθηκεύει κανεί όλο ένα και μικρότερα δεδομένα και ουσιαστικά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται εκεί που παράγονται, διότι θα παράγουμε τόσο πολλά δεδομένα που θα κοστίζει τρομακτικά και θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και ενεργοβόρο το να αποθηκεύσει κανεί όλα αυτά τα δεδομένα. Ε, οπότε θα τα χρησιμοποιεί κανεί και θα τα χάνει με το connected driving, με την ε, συνδεδεμένη οδήγηση για παράδειγμα. Θα υπάρχουν τα δεδομένα διαθέσιμα, αλλά δεν θέλει να τα αποθηκεύεις γιατί πού θα τα αποθηκεύσει. Θα ήταν τεράστιο η ποσότητα. Ευχαριστώ, πολύ. Ε, Thank you so much. κύριος Λαγκοντίνσκι, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηγόντων έστω και καθυστερημένα προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε εσείς την ηγεσία σε αυτό το θέμα. Um, uh, three, very brief. Και σας υποστηρίζω πάρα πολύ. Έχω μερικές σύντομες ερωτήσεις. Κάτι στο οποίο δεν αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας είναι είναι ποιος θα έχει πρόσβαση. Οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση. Σας έχει απασχολήσει αυτό. Το θεωρείτε σκόπιμο ή χρήσιμο γιατί διαφέρουν οι εμπειρογνώμονες. Ε, θα λύσει το πρόβλημα δηλαδή ε, είναι ε, πλήρη στη διαφάνεια ως προς τους κώδικες. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Και επίσης τι θεωρείτε υψηλός κίνδυνος, γιατί και εκεί γίνεται συζήτηση. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων και ανησυχούμε λίγο εμείς ότι υψηλό κίνδυνο θα έχει ένα ορισμό πάρα πολύ τεχνικό, άρα και πολύ μινιμαλιστικό. Εσείς ποια κριτήρια χρησιμοποιείτε μέχρι τώρα στη Λευκή Βίβλο για να ορίσετε τι θα πρέπει να θεωρείτε υψηλό κίνδυνος. Πολύ καλές ερωτήσεις, αλλά και πάρα πολύ ε, δύσκολα θέματα αυτά. Το, ε, η εξηγησιμότητα τι είναι, είναι ζητάς από την τεχνολογία να σου εξηγήσει την τεχνολογία για να μπορείς να παρακολουθείς τι συμβαίνει και πώς αλληλεπιδρούν εκεί οι λογάριθμοι ε, καθώς τρέχουν. Εγώ έχω μεγάλες ελπίδες ότι τελικά θα καταλήξουμε σε κάτι και να υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι που θα φέρουν την τελική ευθύνη. Πολύ συχνά και σε θέματα ανταγωνισμού το λέω. Πώς θα βεβαιωθείς ότι το αλγοριθμό σου έχει σπουδάσει νομική και ξέρει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει και τι πρέπει να αρνηθούν ή αν θέλουν κάτι να αγοράσουν αλλά ε, είναι ε, ένα καρτέλ απέναντι ε, και πώς θα σου πει ο λογαριθμός ότι κοίτα αυτό είναι απέναντι στον ανταγωνισμό. Τώρα αν έχουν οι δημόσιες αρχές πρόσβαση δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν πιστεύω καθόλου ότι μπορούμε να το αναμένουμε από κάθε κράτος μέλος, διότι αυτό χρειάζεται πάρα πολύ ε, εξειδικευμένο προσωπικό και με υψηλές δεξιότητες. Βεβαίως υπάρχει και μια προφανής προσδοκία η τεχνολογία να μην έχει αρνητική επίπτωση η τεχνολογία. Ένα καθρέφτη είναι και τίποτα άλλο. Μας δείχνει τον κόσμο όπως έχει. Παίρνει τα δεδομένα, τα συνθέτει και σου βγάζει το είδωλο του κόσμου που βλέπει ο καθρέφτης αυτός. Στην πρόσληψη, πολλές φορές στο γενικό διευθυντό, το πρώτο κριτήριο, ας πούμε, είναι να είναι άνδρας. Γιατί στα δεδομένα βλέπει ο λογάριθμος ότι όσοι προσλαμβάνουν γενικού διευθυντέ, εκτελεστικούς διευθυντέ, προτιμούν άνδρες, αλλά θα το βάλει πρώτο κριτήριο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τεχνολογία τόσο πολύ, αλλά με τα χρήματα. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις ορχήστες. Όταν άρχισαν ε, ε, να ε, προσλαμβάνουν κόσμο με ακροάσεις πίσω από μια κουρτίνα που δεν έβλεπαν τον υποψήφιο, ε, έσπασε αυτή η προκατάληψη και έσπασε και η διάκριση του φίλου. Το πώς θα είναι ουδέτερη δηλαδή και η τεχνολογία. Και το άλλο ερώτημά σας για τον υψηλό κίνδυνο. Μπορεί κάτι σε μια εφαρμογή να είναι υψηλός κίνδυνος και σε μια άλλη να είναι χαμηλός κίνδυνος. Και δύο εφαρμογές χαμηλού κινδύνου ενδεχομένως όταν συνεργάζονται μπορεί να δίνουν υψηλό κίνδυνο. Εξαρτάται από τον κλάδο και από τη συμμετοχή των ανθρώπων. Ας πούμε, στο τηλέφωνο σας, αν έχετε ένα αυτόματο μεταφραστή και δεν τα λέει πολύ καλά, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις ένα λογισμικό για πυροτεχνήματα, α πούμε, που δεν τα εξαγεί καλά, είναι πολύ διαφορετικό το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο, αλλά πώς να γίνει διάκριση στις γκρίζε ζώνες, που δεν είναι και πολύ, μόνο γκρίζα ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο, είναι πολλά τα χρώματα. Και ακριβώ επειδή είναι τόσο λεπτές οι διαφορές και τα κριτήρια, πολλά εξαρτώνται από την εφαρμογή την ίδια. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπράιερ. Ευχαριστώ, κύριε Βεστάγκερ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, σας ευχαριστώ και για την ειλικρίνειά σας, για τη συζήτηση εδώ μαζί μας, για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες για την ομάδα υψηλού επίπεδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ποντάρει πάρα πολύ στη βιομηχανία εκεί και κυριαρχεί η βιομηχανία. Εγώ θα επιθυμούσα να είναι διαφορετική η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τη συγκεκριμένη πολιτική υπάρχουν κάποιες απαιτήσει διαφάνειας κτλ. Και πώς χρησιμοποιούμε και εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει αυτό να συνοδεύεται και από κόκκινες γραμμές και περιορισμούς που δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αναφερθήκατε ε, σε μια υπόθεση που είναι η αναγνώριση των ε, χαρακτηριστικών του ε, προσώπου. Διέρευσε όμως κάτι στο πολίτικο, γιατί γενικά με την αναγνώριση των χαρακτηριστικών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Μπορεί να υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος, σε δημόσιους χώρους, ένα πλήθος ε, ανθρώπων που αυτό είναι διαφορετικό από το να χρησιμοποιείς ε, την ε, αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου κάποιων που καταζητείται, ας πούμε, που ένα ένταλμα. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα μορατόριο. Αυτό το ζητούμε για κάθε είδους μαζική παρακολούθηση του πληθυσμού και στο συγκεκριμένο. Να μην χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση των προσώπων σε πλήθη. Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό να περιοριστεί σε ανώνυμα δεδομένα. Να μην ξανανοίξει το θέμα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Στη Λευκή Βίβλο. Το αντίθετο θα πρέπει να συζητήσουμε πώς πρέπει να επεκταθεί αυτός ο γενικός κανονισμός, διότι μέχρι στιγμής περιορίζεται σε αλγορίθμους που παίρνουν αποφάσεις. Μα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τις παίρνουν οι αλγόριθμοι τις αποφάσεις, αλλά τις καθορίζουν ή τις υποστηρίζουν ή τις καθοδηγούν ανάλογα με το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουν. Αυτό καθόλου δεν το εξετάζει ο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι στιγμή. Μήπω λοιπόν επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή του. Και τέλο, για τι ψηφιακέ υπηρεσίε και τη σχετική νομοθεσία. Τι γίνεται με τη διασυνδεσιμότητα. Υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο και ανταγωνισμό όπως το γνωρίζετε. Και όχι μόνο στα social media και υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων. Υπάρχουν μεγάλα μονοπόλια. Γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικοί πάροχοι. Και να σας δώσω και μια γεύση της γενικής μας προσέγγισης ε, της κείμενης διατάξης. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προλαμβάνετε ιδιωτική λογοκρισία ή ενδιάμεση δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε τέτοιου είδους λογοκρισίας με φίλτρα ή ακόμα και η ιδιωτική αστυνόμευση. Θέλουμε να αποφασίζουν ανεξάρτητες δημόσιες αρχές για αυτά τα πράγματα. Θα γνωρίζετε τη θέση του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό, για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Νομίζω προς τα εκεί θα πρέπει να στραφεί και η γενικότερη πολιτική. Um, I'm είπαμε, ένας θέμα ρωτάει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνει μόνο μία ερώτηση, ξέρετε. Λέει πως την κυρία Βεστάγκερ πρόεδρος. Βεστάγκερ να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Ναι, καλά τα λέτε. Για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων είχα ασχοληθεί με τη συγκρότησή τους και αυτές οι επτάρχες είναι χρήσιμες. Τα δοκιμάσαμε. Είχαμε 350 αποκρίσεις με όλα αυτά τα ενδελεχή ερωτηματολόγια για τις επτάρχες. Αυτό δούμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν να ε, χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Γιατί έχουμε την πολιτική, στην Κομισιόν και από την άλλη έχουμε τις επιχειρήσεις που στείλουν τα πόδια, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση με πόρους Όποτε και δεν πάει μακριά το θέμα αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Μόνο αν υπάρχει επομένω η εμπιστοσύνη, μόνο κανεί αν το έχει χωνέψει, αυτό το μια επιχείρηση το έχει ε, χωνέψει και να το εμπιστεύεται. Προχωράει. Το θέμα για την επίμαχη τεχνολογία είναι η αναγνώριση προσώπου αλλά και άλλα τα, και τα βιομετρικά. Αυτά θέλουμε να συζητηθούν. Σωστά το είπατε. Έχουμε και εκτεταμένη χρήση και ατομική. Αυτό πρέπει να συζητηθεί. Έγινε και το τεστ στη ΣΥΠΑ. Δύσκολο να δούμε αν απέδωσε η χρήση από την αστυνομία. Τέλο πάντων, στο μέλλον και με την Λευκή Βίβλο θα το συζητήσουμε περισσότερο. Τώρα για την πρόσβαση στα δεδομένα. Ε, βέβαια. Ε, θεωρούμε ότι ο GDPR θα συνεχίσει να ισχύει, δεν θα παρακαμφθεί. Οπότε θα ισχύουν παράλληλα οι ρυθμίσεις. Όποτε γίνεται. Ο πλευράς τεχνικής. έχουμε προσωπικά δεδομένα, δεδομένα που είναι οριακού χαρακτήρα. Εντοπίζουμε κάποιον, έτσι κι τον έχουμε καλύψει, δεν τον ξαναεντοπίζουμε. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχουν περισσότερες προτεραιότητες. Είπαμε πρώτα-πρώτα τα πιο σημαντικά, πρώτα-πρώτα να φροντίσουμε για την υλοποίηση και νομίζω ότι πολλοί οι πολίτες νιώθουν αυτή την αμηχανία, την απογοήτευση, προσπαθούμε να οργανωθούμε στις ρυθμίσεις για να εξασφαλίσουμε ότι το gadget δουλεύει οπότε ακόμα και με τα δικαιώματά μου να προστατεύονται τα δεδομένα. Νομίζω ότι το θέμα καλύπτεται από τις αρμόδιες αρχές διασυνδεθιμότητα, διαλειτουργικότητα για μένα αυτά είναι κορυφές προτεραιότητες είναι θέμα ανταγωνισμού για πολλούς τομείς θα ασχοληθούμε με αυτό. Και με το δίκαιο ανταγωνισμού, με τα δικά μέσα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κυρίως να κάνουμε τους καινούργιους στην αγορά. Και έτσι όμως το πάμε καλύτερα. Οπότε αν δεν το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Με έχετε εντυπωσιάσει. Άλλοι τέσσερις όμως έχουν δει στο λόγο και έχουμε άλλα 15 λεπτά που θα έχουμε τους διερμηνείς κοντά μας. Κύριε Σέσνη. Ποιος? Sorry, Mr. Sejourné. Ο κύριο Σεζουγνέ. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα το όνομά μου. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριο Σεζουγνέ. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ πλήρη εισαγωγή. Η Ευρωπαϊκή Μάλλον, εμείς έχουμε θέματα δεοντολογίας, αστικής ευθύνης ε, και λοιπά στην Επιτροπή μας και στην πνευματική ιδιοκτησία και αυτό το συζητούν οι πολιτικές ομάδες μας. Ποια είναι η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, ε, βιομηχανίας και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας που εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να χαράξουμε, ευρωπαίοι νομοθέτες. Όλοι μου οι συνάδελφοι έκαναν πολλές ερωτήσεις και κάλυψαν όλο το πεδίο. Θέλω να επανέλθω λίγο στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Ε, διέρευσε ένα κείμενο και ε, δημιουργείται τώρα μια συζήτηση γύρω από το moratorium. Αυτό το δίκαιο στάσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέση γι' αυτό και ποια είναι. Μπορείτε να μας τη διευκρινίσετε. Και κάτι άλλο έτσι προς διερεύνηση που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν συζητείτε, αλλά είναι το θέμα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των προσωπικών ιδιωτικών δεδομένων. Τι θα κάνουμε τώρα, αγορά δεδομένων. Κάθε χρήστη έχει δικαίωμα να πουλάει τα δεδομένα του, άρα και δικαίωμα να μην τα πουλάει. Ε, αυτό το έχετε σκεφτεί καθόλου ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ενδεχομένω πρέπει να το διερευνήσουμε στο Κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Uh, uh, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τη διατύπωση στη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε δεν μπορώ να σας πω πώς ακριβώς θα διατυπωθεί. Αλλά η προσέγγιση για τις ευαίσθητες όπως τις ονομάζουμε τεχνολογίες ή τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία σίγουρα θα είναι πολύ προσεκτική. Έτσι θα εφαρμόσουμε στην πραγματική ζωή τις αξίες μας. Το ότι δεν θα υπόκειται ο καθένας μας σε οποιοδήποτε είδους παρακολούθηση. Και ελπίζω ότι θα γίνει μια ευρύτατη συζήτηση που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική και όπως προείπα αυτό δεν αφορά μόνο την παρακολουθήση σε δημόσιους χώρους αλλά και διάφορες άλλες ε, χρήσεις ε, σε αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο στο πλαίσιο μιας αστυνομικής ε, Επιχείρηση ε, στα σύνορα, πώς μπορούμε δηλαδή να διασφαλίσουμε και βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα η ηθική, μα, ε, μας, οι αξίες μας, ε, τα πρότυπά μας πρέπει να εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή. Πιστεύω ότι σε κάποιους τομείς οι τεχνολογίες αυτές θα αποδειχθούν χρήσιμες. Ωστόσο πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γίνει εκτενή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα και για αυτή τη συζήτηση θα καλέσουμε ειδικού, διότι ξεκινάμε με την πρόποθεση ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι είναι πολύ δύσκολη διαφορετικά η ε, διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών αξιών. Τώρα για την ψηφιακή αγορά. Με απογοητεύει, για να σας το πω καθαρά, η αγορά. Περίμενα ότι μετά από τον GDPR ε, θα υπήρχαν περισσότεροι διαμεσολαβητές που θα παρέχαν οι υπηρεσίες ε, σε πολίτες για τη διαχείριση δεδομένων κτλ. Δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί στο μέλλον αυτή η ιδέα. Υπάρχει και μια άλλη ιδέα που ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Η εξή. Όταν ένα φορολογούμενο δημιουργεί δεδομένα, δηλαδή ένα δημόσιο αγαθό, πώ θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά. Η θέση τη Κομισιόν είναι φυσικά ανοιχτά δεδομένα για όλου. Αλλά καθώς μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου ο όγκος των δεδομένων θα είναι τόσο πολύ μεγαλύτερος και θα είναι πολύ δύσκολο να διατεθούν όλα αυτά τα δεδομένα από τους φορολογούμενους οι οποίοι ε, πληρώθηκαν για αυτό το νέο πόρο για να παρασχεθούν αυτά τα δεδομένα στους επιχειρήσεις. Ουσιαστικά θα υπάρξει μία αγορά δεδομένων. Αυτό είναι το ερώτημα βασικά. Και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και εγώ τις δικές σας απόψεις για αυτό το ζήτημα, διότι είναι κάτι που συζητείτε εδώ και καιρό. Και όσον αφορά την αρχή, τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τους πόρους. Ευχαριστούμε, κύριο Βό. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλές ερωτήσεις, κάποιες ε, τις απαντήσατε ήδη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να λάβω θέση σε κάποια σημεία. Πρώτον, η αναγνώριση προσώπου. Δεν καταλαβαίνω τι πλεονέκτημα υπάρχει όταν πάει κανείς και λέει αποθηκεύουμε, ε, σταματάμε συγγνώμη τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου στην Ευρώπη. Επίσης, ε, μπορεί να στείλουμε έτσι ένα λάθος μήνυμα όσον αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες ότι προσπαθούμε να τις σταματήσουμε διότι προσπαθούμε να τις ξεκινήσουμε, ναι, να τις βάλουμε μπρο, αλλά πάμε να κάνουμε κάτι, αν κάνουμε κάποια προσπάθεια να σταματήσουμε την εξέλιξη, πιστεύω θα ήταν λάθος. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, σε αυτό το τομέα θα έχουμε να κάνουμε ε, πάντα με τον GDPR και θα, ερχόμαστε, θα μας δημιουργεί προβλήματα. Αυτός ο βασικός κανονισμός λοιπόν θα πρέπει να ε, τον χρησιμοποιήσουμε κάποιος δημιουργικά όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες ε, και επίσης και με το πώς ε, θα τον χειριστούμε. Και με την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε, για παράδειγμα, τον καρκίνο. Για αυτό το σκοπό χρειαζόμαστε πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία είναι και ευαίσθητα σύμφωνα με τον κανονισμό. Αν όμως δεν, πάρουμε, δεν λάβουμε αυτά τα δεδομένα, διότι έχουμε πολύ ψηλέ απαιτήσει για την προστασία των δεδομένων, εκ των προτέρων έχουμε χάσει τον ανταγωνισμό σε αυτό το επίπεδο. Οπότε χρειαζόμαστε μια λογική έξυπνη λύση για να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον βασικό κανονισμό προστασίας των δεδομένων σε συνδυασμό με την καινοτομία. Ε, επαναχαρακτηρισμό ενδεχομένως ε, δεδομένων, οτιδήποτε. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε κάποια δημιουργικότητα ώστε να είναι δυνατή καινοτομία και σε αυτόν τον τομέα. Επιπροσθέτως, ε, μια άλλη σκέψη Αφενός ε, θέλουμε να συναγωνιστούμε με τις άλλες ε, περιοχές του κόσμου, Τσίπα, την Κίνα και να μένουμε στο ε, παρόμοιο επίπεδο. Με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα δεν θα λειτουργήσει αυτό. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί μόνο αν η Ευρώπη λειτουργεί ως ε, ένα ενίος φορέας. όχι δηλαδή μόνο η Γερμανία να υπερασπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δικά της συμφέροντα και η Γαλλία τα δικά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ε, υπερασπιζόμαστε το ε, ευρωπαϊκά συμφέροντα, πράγματα που να μπορούμε και αποτελεσματικά να εφαρμόσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή να αλλάξουμε νοοτροπία. Εάν δεν καταφέρνουμε δηλαδή η Ευρώπη να υπερασπίζεται το συμφέροντά της ως ένας φορέας, μόνο έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε παγκοσμίω. Και εκεί τίθε το ερώτημα. Θέλουμε πραγματικά ψηφιακή εσωτερική αγορά. Αν ναι, τι νομικό πλαίσιο θα χρησιμοποιήσουμε, τι νομικό εργαλείο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε, θέλουμε πλήρω εναρμονισμένη εσωτερική ψηφιακή αγορά. Διότι για μένα αυτό θα σήμαινε και κανονισμούς. Ξέρω ότι είναι δύσκολο με τα κράτη-μέλη διότι παντού υπάρχουν εθνικά συμφέροντα, εθνικά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι εάν δεν υπερβούμε αυτό το πρόσκομα, η εσωτερική αγορά θα παραμείνει κατακρεματισμένη για πάντα. Οπότε πρέπει να κάνουμε και αυτό το βήμα. Και μετά μια τελευταία ιδέα. Είναι και θέμα έκφρασης εδώ, του πώς θα το πούμε δηλαδή. Εδώ, αν θέλουμε να παραμείνουμε ε, στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες περιοχές του κόσμου, έχουμε διαθέσει και τα οικονομικά μέσα, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις για το πολιτισμό-οικονομικό πλαίσιο έχουμε ορίσει τις σωστές προτεραιότητες και για τον ψηφιακό τομέα. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι η μόχλευση που θέλουμε να επιτύχουμε αυτή τη στιγμή με την Πράσινη Συμφωνία και που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε και με την ψηφιοποίηση, ε, δεν ξέρω μήπως είναι σωστή αυτή η μόχλευση, μήπως μέχρι στιγμή ε, δεν, δεν έχουν παρασχεθεί επαρκή μέσα στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, και εκεί φυσικά υπάρχουν δυσκολίε και με τα κράτη-μέλη, αλλά πιστεύω ότι τώρα έχει έρθει η χρονική στιγμή, είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να πούμε ότι μάλλον πρέπει να το προσεγγίσουμε διαφορετικά. Και όσον αφορά δηλαδή τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά, να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ε, λάβει, έχουμε ορίσει τι σωστέ κατευθύνσει. Um, έχετε δίκιο ότι ο κόσμος ε, συνεχίζει να προχωράει γύρω μας, αλλά αλλάζει κιόλας. Και όλες οι κοινοτομίε δεν καταλήγουν σε κοινωνίες που θα θέλαμε να ζούμε σε αυτές. Και στην Ευρώπη οι εκπρόσωποι μας στις δημοκρατίες μας πάντα τραβούσαν γραμμές ότι αυτό το κάνουμε το άλλο δεν το κάνουμε. Ας πούμε οι αγρότες στην πλειονότητά τους ε, προσέχουν πάρα πολύ πώς χρησιμοποιούνται ε, πώς χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα ε, και προσέχουν και τα ζώα τους. Αλλά δεν μπαίνουμε στο κίνδυνο και στην περιπέτεια να μας μολύνουν το νερό, το πόσιμο όσοι δεν τα χρησιμοποιούν με σύνεση. Γι' αυτό νομοθετούμε. Ας πούμε τι κάνουμε με τα ζώα, τα κτηνοτροφικά και το πόσιμο νερό. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τρόπος εργασίας. Οι δημοκρατίες βάζουν το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο και εντός αυτού εργάζονται οι υπηρεσίες, οι πολίτες και η αγορά. Ε, είναι όμως πολύ θεμητό να πούμε ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο και να μπορούν εκεί μέσα οι πολίτες να ζεστάνονται άνετα μέσα στις κοινωνίες τους. Και σε αυτό έχουμε καταλήξει μετά από ατέρμονες συζητήσεις και τελικά νομοθετούμε και αυτό ισχύει ως ε, δίκαιο. Βέβαια μπορούμε πάντα να συζητούμε πού γίνεται έρευνα, πού σταματάει η έρευνα, τι ε, είναι ατελέσφορο αλλά ε, πρέπει να γνωρίζουμε πώς ε, λειτουργούν αυτές οι τεχνολογίες, ε, οι πάρα πολύ ευαίσθητες, πώς τις χειρίζεσαι και θα πρέπει ο κόσμος να εμπιστεύεται την κοινωνία. Και σιγά σιγά πέφτει η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στην τεχνολογία. Όχι για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επειδή κυκλοφορούν διάφορες φωτογραφίες ως μειόφυλαν ή κάποιο σου στέλνει ένα mail ότι θα σου στείλει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γυναίκε είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Όλα αυτά δημιουργούν μια δυσφορία στον κόσμο. Σου λέει δεν θέλω αυτή τη τεχνολογία. Ε, ε, εμείς πρώτα δείχνουμε με την τεχνολογία τι μπορούμε να κάνουμε και μετά πρέπει να δημιουργήσουμε και την εμπιστοσύνη σε αυτήν. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων να έχουμε ένα σωστό πλαίσιο. Έχουμε μια συντηρητική προσέγγιση. Θα πρέπει να συνεργαστούν οι διάφοροι επαγγελματίε τώρα για να δουν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Έχετε απολύτως δίκιο λέγοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει θαύματα εάν συμφωνήσει ε, δεν υπάρχει σχεδόν ε, κάτι αδύνατο. Και πρέπει να συμφωνήσουμε και για τον προπολογισμό όμως, γιατί χωρίς χρήματα ό,τι ιδέες και να έχουμε, τι να τις κάνουμε. Αλλά και με την καλύτερη χρηματοδότηση, που ακόμα δεν έχω απεμπολίσει τις ελπίδες μου, θα πρέπει να οργανώσουμε την έρευνά μας και την καινοτομία μας. Αλλιώς δεν πρόκειται να φτάσουμε τα παγκόσμια επίπεδα, ούτε να δημιουργήσουμε αυτό το οικοσύστημα που σας είπα, όπου το ταλέντο προσελκύει ταλέντο για να παραμείνει στην Ευρώπη και ε, να υλοποιηθούν κάποια από αυτά τα πράγματα. Αλλά θα αποτύχει το πείραμα. Αν δεν έχουμε τα χρήματα, όσες καλές ιδέες και να έχουμε, θα πάνε στο βρόντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κάρεν και μετά ο Τίμο Βέλκεν τελευταίος. Η κυρία Μέλχιορ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και που τα συζητάτε και ελπίζουμε να συνεχιστεί η επαφή μας από του χρόνου. Έχουμε αυτούς τους εμπειρογνώμονες που είπατε ήδη έχουν παράσχει συμβουλές χρήσιμες και για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς διαφέρει αυτή και η νομοθεσία της σε σχέση με την νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τα είπατε στην εισήγησή σας όσον αφορά την αριστεία και την εμπιστοσύνη. Μπράβο. Αλλά αυτά πώς εφαρμόζονται στις πλατφόρμες μέσω ενημέρωσης και στα θέματα κρυπτογράφησης και κωδικοποίησης. Είναι θέμα για ασφάλειες, όχι μόνο εμπιστοσύνης. Να μην έχουμε διαρροές δεδομένων, οπότε πάει η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά ε, την αριστεία. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Δεν θα πρέπει να έχουμε εκεί χειραγωγήσει από κάποιου αλγορίθμου εκτό ελέγχου. Υποχρέωση λογοδοσία ε, και διαφάνεια κλπ. Όλα αυτά χρειάζονται όσον αυτό το γίγνεσθε. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά στη ζήμωση γιατί το τι θα κάνουμε με την ε, την νομοσύνη και την νομοθεσία για τα ψηφιακά σας το λέω γιατί τελικά είναι θέμα κώδικα τι θα κάνουμε πώς, πώς έχουμε να καλύψουμε με αυτή την νομοθεσία την τεχνητή νομοσύνη Ευχαριστούμε που μας έδωσαν παράταση οι διερμηνείς. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει άλλη μία ερώτηση. Η Επίτροπος. Ξέρω, ξέρω ότι μακρηγορώ ε, στις απαντήσεις. Εγώ φταίω για αυτό που είπατε πάντως. Για να δούμε. Τι, τι μας είπατε. Μια που για μένα ένα παράδοξο είναι ότι στα ψηφιακά. Δεχόμαστε πράγματα που δεν δεχόμαστε στον πραγματικό κόσμο. Ήρθε όμω η ώρα να βγούμε από αυτό το όνειρο ότι το ίντερνετ είναι χώρος ελευθερίας και ανάπτυξης προσωπικότητας. Άλλος κόσμος είναι που τον δημιουργήσαμε σε αυτό τον ψηφιακό χώρο. Ίσως αυτά όλα ισχύανε στην αρχή-αρχή.